Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 10 marca Λοιπόν, είχε διακοπεί στις 10 Μαρτίου του 2011 η Σύνοδος και συνεχίζεται σήμερα. Τα πρακτικά και το κείμενο για τη Σύνοδο της 10ης Μαρτίου του 2011 έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν τυχόν σχόλια. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, οπότε θεωρούνται τα πρακτικά ως ε, εγκεκριμένα. Λοιπόν, τώρα κάποια σχόλια στην αρχή της ε, συνεδριάσεώς μας θα ήθελα να καλωσορίσω τη Μαρία Ρωμάνα Ντεκάσπαρη, τη θηγατέρα του μεγάλου ηγέτου Αλτσίντε Ντεκάσπαρη, που ήταν ένας από τους ιδρυτές πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Δεύτερη πληροφορία που έχω να σας δώσω. Ανησυχητικά νέα λαμβάνουμε από γειτονικέ χώρες Μπαχρέιν, Συρία και Ιεμένη. Σε όλες αυτές τις χώρες οι διαδηλώσεις κατεστάλησαν ε, και ήταν άνθρωποι αυτοί που διαδήλωναν για περισσότερη δημοκρατία. Και